Meine sehr geehrten Damen und Αξιότιμοι και κύριοι. Μεγαλειότατε. Εξ ονόματος των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σας καλωσορίζω θερμά στο Στρασβούργο, στο Κοινοβούλιο. Είναι η τέταρτη επίσκεψή σας στο σώμα και δείχνει πόσο εκτιμάτε, πόσο εμπιστεύεστε και πόση φιλία αισθάνεστε έναντι του σώματος αλλά και των πολιτών, άνδρων και γυναικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Καλωσορίζω και τα μέλη της αντιπροσωπείας σας, ιδιαιτέρως τους προέδρους των δύο κοινοβουλευτικών σωμάτων του Ιορδανικού Κοινοβουλίου, τον φίλο πρόεδρο της Γερουσίας και της Βουλής των του Σώματος των Βουλευτών, της Βουλής των Εκπροσώπων. Ιδιαιτέρως δε με χαρά καλωσορίζω τους φοιτητές από την Ιορδανία, φοιτήτρες και φοιτητές που έχετε φέρει μέσα στην αντιπροσωπεία σας. Σας καλωσορίζουμε όλους θερμά. Μεγαλειότατε εξ ονόματος του Κοινοβουλίου επαναλαμβάνω τα λόγια που ακούσατε νωρίτερα που οφείλω όμως να επαναλάβω και την παρουσία σας. Εκφράζουμε τα βαθύτατα συλληπιτήριά μας, τη θλίψη μας για τον αποτρόπαιο θάνατο το Μουάς Καζασπή, πιλότου της πολεμικής αεροπορίας, της βασιλικής Ιορδανικής αεροπορίας. Οι σκέψεις μας και τα συλληπιτήριά μας με την οικογένειά του και του οικείους του. Ο αποτροπιασμός από την ανακοίνωση αυτής της φρικτής είδηση και τις εικόνες του σκληρού αυτού θανάτου, του πιλότου σας, ξεπερνούν την ε, ανθρώπινη φαντασία. Πώς μπορεί κανείς δηλαδή να διαπράττει τέτοιες πράξεις. Πρόκειται για πράξεις εγκληματικές και βάρβαρες του Ισλαμικού λεγόμενου κράτους που μας γεμίζουν με αποτροπιασμό, που έρχονται αντίθετες με οποιαδήποτε αξία και αρχή μας ενώνουν. Η Συρία έχει δει να φεύγουν για να γλιτώσουν από τον εμφύλιο πόλεμο και, τον αποτρόπαιο, και τις αποτρόπαιες πράξεις του Ισλαμικού κράτους εκατοντάδες χιλιάδες πολιτών της που βρήκαν ζεστή υποδοχή στην πατρίδα σας, στην Ιορδανία από τον Ιορδανικό λαό. Ξέρουμε πόσο μεγάλες είναι οι προκλήσεις ενώπιον των οποίων βρίσκεστε. Επιτρέψτε μου λοιπόν, εξ του Κοινοβουλίου, να εκφράσω σε εσά και τον λαό σας, άλλωστε το δείχνουν και τα ε, χειροκροτήματα, την αλληλεγγύη μας και την υποστήριξή μας σε αυτή την προσπάθεια. Θέλουμε να προχωρήσει και να υποστηρίξουμε την Ιορδανία στο δρόμο για τις πολιτικές μεταρρυθμίσεις και τις οικονομικές μεταρρυθμίσεις που εσείς ε, ξεκινήσατε μεγαλειότατε και που αποτελούν επιθυμία του λαού σας. Αυτό ανταποκριθήκατε, γιατί αναγνωρίσατε ότι οι μεταρρυθμίσεις, η ειρήνη, ο σεβασμός των ανθρωπινών ε, οι μεταρρυθμίσεις θα μπορούσαν να φέρουν την ειρήνη και το σεβασμό των ανθρωπινών δικαιωμάτων στη χώρα σας και την περιοχή. Συμμετέχετε επίσης ε, στη Μεγάλη Διεθνή Συμμαχία κατά του λεγόμενου Ισλαμικού κράτους. Σε αυτή είναι εταίροι η Ιορδανία και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Θέλουμε ο Ιορδανικός λαός να ζει σε όρους αξιοπρέπειας, μέσα σε ένα ασφαλές περιβάλλον. Αυτό το εξασφαλίσετε εσείς μεγαλότατα εδώ και πολλά χρόνια, συμβάλλοντας σημαντικά στην διασφάλιση και την επάνωδο της ασφάλειας στην περιοχή σας. Είναι ηγετική η στάση της χώρας σας και η αντίσταση που προβάλλει στις προσπάθειες να διεισδύσουν ακραίοι και τρομοκράτες. Σε αυτό οφείλουμε να επιδείξουμε το μέγιστο σεβασμό μας. Έχετε επιδείξει σε δύσκολη περίοδο πολύ μεγάλο σεβασμό στις μειονότητες και διαλλακτικότητα ως κράτος με τη δυνατότητα που εξασφαλίζεται σε, διαφορετικούς, σε λαούς από διαφορετικές προελεύσεις και θρησκείες να συμβιώνουν ειρηνικά. Εξού και ήταν πολύ σημαντικό σημάδι η παρουσία σας στην ε, διαδήλωση που έγινε μετά τις τρομοκρατικές επιθέσεις στο Παρίσι και το περιοδικό Σαρλί Εμπτό, για την οποία και σας ευχαριστώ θερμότατα εκ μέρους του Κοινοβουλίου. Ένα σημάδι λοιπόν, ένα μήνυμα με το οποίο δείξατε ότι η Ορδανία θα κάνει ακόμη περισσότερα κατά της τρομοκρατίας και υπέρ της διαλλακτικότητας και της ειρήνης. Και επίσης, επιτρέψτε μου ολοκληρώνοντας, να χαιρετήσω την ακαταπώνητη στράτευσή σας και προσήλωσή σας στην επίλυση ειρηνικά της Ισραηλοπαλαιστινιακής διένεξης. Σας το είπα και κατηδίαν. Είναι ένας αγώνας τον οποίο και εμείς συμμεριζόμαστε και δεν θέλουμε να, ε, να διακοπούν οι προσπάθειες για την ειρηνική επίλυση του προβλήματος αυτού. Τους αληθινούς φίλους τους βλέπει κανείς στις δύσκολες ε, περιόδους. Εμείς οι Ευρωπαίοι θεωρούμε ότι είναι πραγματικός φίλος ο Ιορδανικός λαός και ο βασιλεύς του. Καλώς ήρθατε. Σας χαιρετίζω θερμά και σας δίνω το λόγο. Κύριε Πρόεδρε, αξιότιμοι βουλευτές. Σας ευχαριστώ θερμά. Η Ορδανία θεωρεί πολύτιμους ε, τους μακροχρόνιους ε, δεσμούς φιλίας που τη συνδέουν με το μεγάλο αυτό θεσμό. Και σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση που μου απευθύνεται να μιλήσω εδώ σήμερα. Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω τους πολίτες της πόλης του Στρασβούργου για την θερμή τους φιλοξενία. Η πόλη αυτή πάντοτε αντιπροσωπεύει το σύμβολο της μετάβασης από τον πόλεμο στην ειρήνη. Είναι ένα σύμβολο της συμφιλίωσης και της ενότητας της Ευρώπης. My Αγαπητοί φίλοι, οι λαοί ανθούν όπου υπάρχει αμοιβαίος σεβασμός. Ε, πάνω σε αυτόν τον αλληλοσεβασμό άλλωστε βασίζεται ο πολιτισμός ε, και έτσι θα έχουμε ένα καλύτερο μέλλον. Όμως η συνύπαρξη είναι κάτι που πρέπει να το κερδίζει η κάθε γενιά ξανά και ξανά. Το κοινό καλό μπορεί να το υπερασπιστούμε μόνο αν επαγρυπνούμε και αν αναλαμβάνουμε δράση και αυτό δεν σημαίνει μόνο μέτρα ασφαλείας. Θα πρέπει η ανθρωπότητα να εξοπλιστεί με ιδέες, με δικαιοσύνη και με οικονομική και κοινωνική ένταξη. Σήμερα οι προκλήσεις αυτές έχουν μια ιδιαίτερη σημασία ο κόσμος μας αντιμετωπίζει την επίθεση τρομοκρατών που χαρακτηρίζονται από μια αδίστακτη φιλοδοξία. Κίνητρό τους δεν είναι η πίστη, είναι η ισχύς, η δύναμη την οποία προσπαθούν να αποκτήσουν ε, ξεσκίζοντας χώρες και κοινότητες ε, σε μυσαλόδοξες ε, συγκρούσεις και με βία και οδύνη σε όλο τον κόσμο. Η στιγερή δολοφονία από τον Ντάεσ, το Ισλαμικό κράτος του Ιορδανού ήρωα πιλότου είναι κάτι το οποίο γέμισε αγανάκτηση όλους τους Ιορδανούς και αποτροπιασμό όλου τον κόσμο. Ήταν γρήγορη, σοβαρή και αποφασιστική η αντίδραση της Ιορδανίας και ο αγώνας μας θα συνεχιστεί. τόσο εμείς ε, όσο και άλλα αραβικά ε, και μουσουλμανικά κράτη περασπιζόμαστε όχι μόνο το λαό μας αλλά και την πίστη μας. Πρόκειται για έναν αγώνα που θα πρέπει να τον διεξάγουν πρώτα απ' όλα τα μουσουλμανικά έθνη. Είναι ένας αγώνας που πρέπει να δοθεί εντός του Ισλάμ. Ταυτόχρονα να όμως ο κίνδυνος του εξτρεμισμού πρέπει να γίνει αντιληπτός για αυτό που πραγματικά είναι. Είναι ένας παγκόσμιος κίνδυνος. Η απειλή δεν εντοπίζεται μόνο στη Συρία και το Ιράκ. Έχει χτυπήσει τη Λιβύη, την Ιεμένη, το Σινά, το Μαλί, την Ιγυρία, το κέρας της Αφρικής, την Ασία, την Αμερικανική Ήπειρο και την Αυστραλία. Η Ευρώπη επίσης έχει υποστεί ποτρόπες ε, επιθέσεις και έδειξε επίσης αδάμαστο σθένος. Οι φίλοι σας είναι μαζί σας. Τον Ιανουάριο η Ράνια και εγώ μαζί με εκατομμύρια ανθρώπους στη Γαλλία περπατήσαμε, διαδηλώσαμε από κοινού ενωμένοι κατά της βίας και του εκφοβισμού. Αγαπητοί φίλοι, Υπάρχουν άνθρωποι που ζουν σήμερα στην Ευρώπη και θυμούνται τα δεινά ε, που έπληξαν την Ήπειρο στα τέλη της δεκαετίας του 30 και το παγκόσμιο πόλεμο που ακολούθησε λόγω μιας επιθετικής, επικτατικής ιδεολογίας που ήταν βασισμένη στο μίσος, ε, και που παραγνώριζε την ίδια την πεμπτουσία της ανθρωπότητας. Αυτός ο πόλεμος στην Ευρώπη έγινε παγκόσμιος πόλεμος. Σήμερα έναν παρόμοιο πόλεμο δίνουμε κι εμείς. Ένα πόλεμο κατά μιας επεκτατικής ιδεολογίας η οποία τρέφεται με μίσος, η οποία διαπράττει δολοφονίες στο όνομα του Θεού και της ε, θρησκείας για να δικαιολογήσει ε, πράξεις ε, κακές που δεν έχουν καμία σχέση με τη θρησκεία. Είναι ένας πόλεμος κατά τρομοκρατών που δεν σέβονται τις αξίες του Ισλάμ και της ανθρωπότητας. Η νίκη εξαρτάται από την ενότητα η δική μας νίκη εξάρτητα από τη δική μας ενότητα και ο ρόλος της Ευρώπης είναι σημαντικός. Μόνο με συνεργασία μπορούμε να κλείσουμε ε, τη στρόφιγγα της ε, υποστήριξης προς τους τρομοκράτες και άρα να τους κάνουμε να χάσουν. Και επίσης είναι πάρα πολύ σημαντικό οι περιοχές μας να ανανεώσουν την πηγή της μεγάλης τους δύναμης που είναι ο αλληλοσεβασμός που μας συνδέει και μας υποστηρίζει και ιδίω η νεολαία. Θα πρέπει να εμπνέεται από τις αξίες οι οποίες απορρίπτουν τη βία, δημιουργούν ειρήνη και κοινωνίες αλληλέγγυες. Θα ήθελα να σας προτείνω τρεις σημαντικούς τομείς. Ο πρώτος ε, είναι μια πραγματική διαθρασκιακή προσέγγιση εκεί που ζει ο καθένας μας. Ε, Διανέργεια ενός διαλόγου ε, βασισμένου στο σεβασμό. Αυτό είναι το λίκνο όλων των κοινωνιών. Η επίθεση, ο αποκλεισμό άλλων, ε, η προσβολή άλλων λαών, τη πίστη του, των πεπιθήσεών του, των του, δεν είναι αυτό ο δρόμο προ τα εμπρό. Το μέλλον έγκυται στην ενότητα και το σεβασμό και όχι στη διέρεση και στα στερεότυπα. Η Ευρώπη είναι ένα σημαντικό εταίρος σε αυτή την προσπάθεια. Ιδίως ε, για να βοηθήσει και να ανακόψει, να βοηθήσει στην ανακόπη μάλλον αυτής ε, της ε, αύξησης της Ισλαμοφοβίας. Είναι ένα δηλητήριο που βασίζεται σε φαλκιδευμένες ιδέες και το αξιοποιούν αυτοί οι εξτρεμιστές. Γι' αυτό και είναι σημαντικό να διευκρινίσουμε τι σημαίνει πραγματικά να είσαι μουσουλμάνος. Και εγώ και αναρρύθμιτοι άλλοι μουσουλμάνοι. Διδαχθήκαμε από την πιο νεαρή μας ηλικία ότι η θρησκεία μας ε, απαιτεί το σεβασμό και την αγάπη για τον πλησίον. Ο προφήτης Μωάμεθ, ε, ειρήνη και ευλογία αυτό, είπε «Κανείς από εσά δεν έχει πίστη εάν δεν επιθυμεί για τον πλησίον του αυτό που επιθυμεί για τον εαυτό του». Αυτό σημαίνει να είσαι μουσουλμάνος. Μεταξύ πολλών ε, επωνυμιών του Θεού ακούμε ο φιλέσπλαχνος, ο πανελέμων Θεός. Κάθε μέρα σε όλη μου τη ζωή έχω ακούσει και έχω χρησιμοποιήσει το χαιρετισμό ασαλάμα λέκουμ που ουσιαστικά είναι μια επιθυμία να είναι ευλογημένη με ειρήνη οι συνανθρωποί μας. Αυτό σημαίνει να είσαι μουσουλμάνος. Πάνω από χίλια χρόνια πριν ε, τι συμβάσει της Γενέβη, οι μουσουλμάνοι στρατιώτες παίρνανε την εντολή, τη διαταγή να μην σκοτώσουν ποτέ ένα παιδί, μια γυναίκα ή έναν ηλικιωμένο. Να μην καταστρέψουν ένα δέντρο, να μην βλάψουν έναν ιερέα, να μην καταστρέψουν μια εκκλησία. Αυτές είναι οι ίδιες αξίες του Ισλάμ, τις οποίες διδαχθήκαμε εμείς ως παιδιά στο σχολείο. Να μην καταστρέφουμε, να βεβηλώνουμε έναν τόπο λατρείας του Θεού. Ούτε τεμένοι, ούτε εκκλησίες, ούτε συναγωγές. Αυτό σημαίνει Αυτό σημαίνει να είσαι μουσουλμάνος. Αυτές είναι οι αξίες που διδάσκω στα παιδιά μου και τις οποίες τα παιδιά μου θα μεταλαμπαδεύσουν στα δικά τους παιδιά. Αγαπητοί φίλοι, είμαι ε, πλήρης αποτροπιασμού και οδύνης από τις πρόσφατες επιθέσεις ε, κατά χριστιανών και μειονοτήτων σε κάποιες χώρες. Πρόκειται για μια επίθεση κατά της ανθρωπότητας και κατά του Ισλάμ. Οι Άραβες χριστιανοί είναι ένα απόσπαστο τμήμα του παρελθόντος, του παρόντος και του μέλλοντος της περιοχής μας. Η Ορδανία είναι μια μουσουλμανική χώρα με μια βαθιά ριζωμένη χριστιανική κοινότητα. Από κοινού ο λαός της αποτελεί μια αδιέρετη κοινωνία. Όλοι είμαστε φίλοι και εταίροι για την οικοδόμηση της χώρας μας. Οι μουσουλμάνοι όλου του κόσμου έχουν ε, έναν πολύ σημαντικό ρόλο να διαδραματίσουν στην παγκόσμια κατανόηση. Όπως και η δική σας έτσι και η δική μας πίστη ζητά έλεος, ειρήνη και ανεκτικότητα όπως και η δική σας προωθεί ε, την ανθρώπινη αξιοπρέπεια, την ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών, γειτόνων, ε, αλλοδαπών, ξένων. Υπάρχουν κάποιοι όμω ε, που είναι εκτό νόμου του Ισλάμ, οι οποίοι απαρνούνται τι αρχέ αυτέ, όμω του ξεπερνούν ο ωκεανό των πιστών, 1,6 δισεκατομμύρια μουσουλμάνους σε ολόκληρο τον κόσμο. Ουσιαστικά αυτοί οι, μουσουλμα... αυτοί οι τρομοκράτες έχουν κάνει τους μουσουλμάνους όλου του κόσμου το μεγαλύτερό του στόχο. Δεν θα τους επιτρέψουμε όμως να πάρουν όμοιρο τη θρησκεία μας και την πίστη μας. Αγαπητοί φίλοι, ο δεύτερος σημαντικός τομέας που είναι πολύ σημαντικός για να υπάρχει αρμονία στον κόσμο είναι ένα διεθνές σύστημα που θα δίνει σε όλους το σεβασμό που επιθυμούν και που αξίζουν. Πανελειμμένως ακούω το ερώτημα γιατί ο κόσμος δεν υπερασπίζεται τα δικαιώματα των Παλαιστινίων. Συνεχώς βλέπουμε να τελματώνει, ε, να παραμένει στάσιμη ειρηνευτική διαδικασία. Θα ήθελα να σας πω πώς φαίνεται στην πραγματικότητα η κατάσταση. Όλο και περισσότεροι επικισμοί από τους Ισραηλινούς, όλο και λιγότερος ε, σεβασμός για τους ε, υποκατοχή Παλαιστινίους. Αυτή η αποτυχία δείχνει, στέλνει ένα κίνδυνο μήνυμα, διαβρώνει την πίστη στο διεθνέ δίκαιο και τη διεθνή κοινότητα. Απειλεί ένα πυλώνα τη παγκόσμια ειρήνη. Μια σύγκρουση όμω που πρέπει να λυθεί με πολιτικά μέσα, όχι με τη βία, όχι με τη ισχύω και έχει δώσει και ένα πολύ μεγάλο όπλο στις πύρους στους εξτρεμιστές αυτή η αποτυχία, διότι εκμεταλλεύονται τις αδικίες και αυτή τη σοβούσα ε, σύραξη για να δημιουργήσουν ουσιαστικά μια νομιμοποίηση για το κίνημά τους και να στρατολογήσουν ξένους μαχητές και από την Ευρώπη και από όλο τον κόσμο. Είναι καιρός λοιπόν να σκεφτούμε το μέλλον και πώς αυτή η συνεχιζόμενη σύγκρουση θα θρέψει, ε, θα δημιουργήσει περισσότερη βία, μίσος και τρόμο σε όλο τον κόσμο. Πώς εμείς μπορούμε να δώσουμε την ιδεολογική μάχη εάν δεν χαράξουμε το δρόμο προς τα εμπρός, προς την ειρήνη μεταξύ Παλαιστινίων Ισραηλινών. Οι χώρες μας ενωμένε πρέπει να δώσουν την όθηση, να χαράξουν το δρόμο προς τα εμπρός, προς μια τελική ε, πλήρη διευθέτηση αυτού του προβλήματος. Κυρίες και κύριοι, μια τρίτη κρίσιμη προσπάθεια είναι η δημιουργία μιας βαθύτερης ελπίδας. Η ριζοσπαστικοποίηση βασίζεται στην οικονομική ανασφάλεια και τον αποκλεισμό. Για να μπορέσουμε να έχουμε πολλούς ε, άλλους με το μέρος μας έναν ειρηνικό κόσμο, θα πρέπει να τους δώσουμε τη δυνατότητα να ζήσουν μια καλή ζωή, να αναπτύξουν το δυναμικό τους. Είναι ένα ισχυρό μήνυμα σεβασμού το να του βοηθήσουμε. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αναγνώρισε τη σημασία τη δημιουργία κοινωνικών και οικονομικών ευκαιριών, καθώ το 2015 το έχει ονομάσει έτος ανάπτυξη Για την Ιορδανία η ανάπτυξη είναι προτεραιότητα και παρά όλε τι περιφερειακέ προκλήσει δεν έχουμε σταματήσει τι προσπάθειε να αντιμετωπίσουμε τι κατεπήγουσε ανάγκε. Τη δημιουργία θέσεων εργασία, τη βελτίωση τη ποιότητα ζωή, με συνεχεί μεταρρυθμίσει και εταιρικέ σχέσει όπω μαζί με εσά και οι αρχές, οι αξίες της Ιορδανίας είναι σημαντικές. Εμείς εκτιμούμε την ε, ισχυρή εταιρική σχέση που έχουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα μέλη αυτής και είμαστε δεσμευμένοι με τη δική σας υποστήριξη να εργαστούμε από κοινού για να πάμε σε ένα ακόμα πιο υψηλό επίπεδο αυτή την εταιρική σχέση. Η Ορδανία επίσης λαμβάνει πολύ σοβαρά υπόψη τις ηθικές της υποχρεώσεις προς τους άλλους. Δεν έχουμε πολλούς πόρους, όμως ε, έχουμε ανοίξει τις αγκάλες και έχουμε υποδεχθεί τους πρόσφυγες ε, που έχουν φύγει από χώρες όπου σοβούν ε, σύραξ περιφερειακές. Η Ορδανία έχει υποδεχθεί χιλιάδες χριστιανούς από το Ιράκ τον τελευταίο χρόνο Έχουμε επίσης παράσχει καταφύγιο σε 1,4 εκατομμύρια πρόσφυγες από τη Συρία, το 20% του πληθυσμού, πάντα μέσα στα τελευταία χρόνια. Ουσιαστικά αυτό αντιστοιχεί στο να έχει υποδεχθεί η Γαλλία όλους τους Βέλγους. Η μικρή μου χώρα πλέον είναι η τρίτη ε, χώρα που υποδέχεται το μεγαλύτερο αριθμό προσφύγων τρίτη και σας ευχαριστώ όλους όσους μας βοηθάτε να φέρουμε σε πέρα στην τεράστια αυτή ευθύνη. Αγαπητοί φίλοι, η υποστήριξή σας στέλνει ένα μήνυμα, όχι μόνο στο δικό μου λαό, αλλά και όλους όσους επιθυμούν να προχωρήσουν με ειρήνη και με τριοπάθεια. Η Ευρώπη είναι μαζί σας. Οι περιοχές μας, οι λαοί μας δεν μπορούν να βρουν καλύτερους εταίρους γείτονες από ότι είναι ο ένας για τον άλλο. ιστορία, γεωγραφία, το μέλλον μας ενώνουν. Ας μην αφήσουμε κανέναν να μας χωρίσει, διότι μαζί μπορούμε να δημιουργήσουμε πυλώνες αλληλοσεβασμού που θα στηρίξουν το κοινό καλό για τις επόμενες γενιές. Σας ευχαριστώ θερμά. Νομίζω το χειροκρότημα το υπέστητε μεγαλειότατα. Δεν ήταν τόσο ε, σύντομο το χειροκρότημα. Από την άλλη όμως σπάνια βλέπουμε να χειροκροτεί κανείς, να χειροκροτούν οι βουλευτές τόση πολύ ώρα και αυτό δείχνει πόσο εκτιμούν τα λόγια σας. Είμαι βέβαιος ότι θα χειροκροτούσαν ακόμη περισσότερο οι συνάδελφοι. Βλέπουμε από τα λόγια σας για την, ε, από την περιγραφή που δώσατε της περιοχής αλλά και από το δικό σας όραμα πως μιλήσατε εκ βάθους καρδιά. Σας ευχαριστώ θερμά.